έγιναν μεγάλες εξελίξεις, απρόσμενες, ρηξικέλευθες λύσεις για τη Συμφωνία για το Κλίμα. Για πρώτη φορά όλα τα κράτη της γης ενώθηκαν στη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος. Το σημαντικό είναι ε, ότι θέλουμε να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς και θέλουμε να περιοριστούμε ζητούμε στο 1,5% αύξηση. Αυτό είναι μια συμφωνία που δείχνει προς το μέλλον γιατί θα θέλουμε να γίνουμε ένας πλανήτης ουδέτερος ως προς το κλίμα που δεν θα επηρεάζει δηλαδή ε, τα αέρια του θερμοκηπίου, δεν θα τα επηρεάζει και δεν θα επηρεάζεται ο πλανήτης από αυτά. Ε, μεγάλη αλλαγή για τον ε, πλανήτη, αν εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα πρέπει να κάνουμε πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας, και την κατανάλωση ενέργειας. Θα δημιουργηθεί και ένας μηχανισμός ο οποίος κάθε πέντε χρόνια θα μας ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις στην εφαρμογή δηλαδή που πάμε καλά και που πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμφωνία αυτή πρέπει να την εφαρμόζει στο εσωτερικό της και προς τα έξω και βεβαίως να τηρεί και να σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη συμφωνία. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν εδώ και πάρα πολύ καιρό για την επιτυχία της διάσκεψης των Παρισίων Θέλω με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω εσάς, ε, Επίτροπε Κανιέτε, για τη συμμετοχή σας στη διάσκεψη. Ξέρουμε ε, πόσο εντατικά εργασθήκατε. Ευχαριστίες και προς ε, το τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Ξέρουμε ότι η Προεδρεύουσα στο Συμβούλιο συνεργάστηκε εντατικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Φιγκέρες, εκτελεστική γραμματέα και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπανκιμούν. Κυρίες και κύριοι, η γαλλική κυβέρνηση ως ε, αμφιτρίων και οργανώτρια της διάσκεψης ε, κάνε πάρα πολλά πράγματα και ε, τον ε, πρόεδρο ε, της διάσκεψης Λοράν Φαβιού στον Υπουργό Εξωτερικών τον ευχαρίστησα προσωπικά και τον προσεκάλεσα να έρθει και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα εδώ ο κ. Φαμπιούς απεδέχθη την πρόσκληση και τον Ιανουάριο θα έρθει για να μας μιλήσει για τα αποτελέσματα της διάσκεψης. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες που παρευρέθησαν στη διάσκεψη και συνέβαλαν στην επιτυχία της. Ένα θερμό ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια. Τα πρακτικά και τα κείμενα της Δευτέρας Δεκεμβρίου υπάρχουν, ε, υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τα πρακτικά αυτά. Τα πρακτικά εγκρίνονται. Κυρίες και κύριοι, προχωρώ στις ανακοινώσεις. Η Νομική Επιτροπή στη συνεδρίαση